Ε, Αγαπητέ συνάδελφε, είναι μεγάλη χαρά να υποδέχομαι σήμερα τον πρόεδρο της Επιτροπής Αφρικανικής Ενότητας, τον Μουσάφα Φάκη Μοχάματ. Είστε ο πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης που έρχεται στην Ολομέλειά μας. Η Αφρική για μας είναι βασική προτεραιότητα. Συμμεριζόμεθα πολλές ε, αξίες μαζί σας, αλλά και πολλές ε, προκλήσεις, δυσκολίες, ασφάλεια, μετανάστευση, ανεργία, κλιματολογικές αλλαγές. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε την στρατηγική εταιρική μας σχέση και να εργαστούμε μαζί ισότιμα για να μπορέσουμε να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις στις ανησυχίες τις οποίες εκφράζουν οι συμπολίτες μας. Χαιρετίζω τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης στην προσπάθεια κατά της τρομοκρατίας. Η προσπάθειά μας αυτή είναι βασική και στο Σαχέλ και στην περιοχή της λίμνης του Τσάβ και στο κέρας της Αφρικής, ακόμα δε και στην ίδια τη Λιβύη. Έχουμε λοιπόν κοινό συμφέρον να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ώρες, να καταπολεμήσουμε το τράφικινγκ, να προλάβουμε την ριζοσπαστικοποίηση. Είναι απαραίτητο επίσης να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες εργασίας για την αφρικανική νεολαία, στην ίδια όμως την Αφρική. Πρέπει να αναπτύξουμε λοιπόν σε επίπεδο διπλωματίας τις οικονομικές μας σχέσεις και να επενδύσουμε περισσότερο και καλύτερα στην Αφρικανική Ήπειρο εκφράζω τη βαθιά μου ανησυχία για την κρίση σε επίπεδο προμήθειας τροφίμων και τον λοιμό που βασανίζει τεράστιες περιοχές στην Αφρική. Αύριο θα συζητήσω με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για αυτήν την ανθρωπιστική κρίση. Είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με τις αφρικανικές χώρες, όπως επίσης και σε επίπεδο θεσμικό, με την αδελφή οργάνωση, την, Αφρικανική, ε, την Επιτροπή Αφρικανικής Ενότητας. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Monsieur le Président, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξοχότητες, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι διότι μου δίνεται μια σημαντική ευκαιρία να πάρω το λόγο ενώπιον της ε, συνέλευσής σας, η οποία εκπροσωπεί τους ευρωπαϊκούς λαούς στην ποικιλομορφία τους για να μιλήσω για την εταιρική σχέση Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ενισχυθεί από το 2000 από την πρώτη σύνοδο κορυφής στο Κάιρο και έχει ανοίξει ε, τα φτερά της μετά από τα πρώτα αυτά αποφασιστικά βήματα. Είμαι πεπισμένος ότι η επόμενη σύνοδος του Νοεμβρίου, η οποία προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή, θα αποτελέσει και ένα νέο βήμα, ένα νέο στάδιο σε αυτή την πορεία που ε, κάνουμε από κοινού για ένα λαμπρό μέλλον για τους λαούς της Ευρώπης και της Αφρικής. Αυτό το ζεύγος Ευρώπη-Αφρική έχει μια όμορφη ιστορία. Έχουμε περάσει από στάδια σκιάς αλλά και φωτός στο παρελθόν. Σήμερα μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι για τη ζωντάνια του ζευγαριού αυτού, για το δυναμισμό αλλά και για τις υποσχέσεις ε, που δίνει το ένα μέλος στο άλλο ε, για έναν ε, έθριο ουρανό και για μελλοντικές θετικές εξελίξεις. Από την μία και από την άλλη πλευρά της Μεσογείου έχουμε την Αίγυπτο, την Ελλάδα, τη Ρώμη, την Καρθαγένη, ε, τη Φινίκη, ε, όλους αυτές τις περιοχές και τους πολιτισμούς που έχουν ε, υφάνει δεσμούς άρρηκτους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο απικισμός κατά τη διάρκεια των 200 ε, ετών που διήρκησε έθεσε τους πολιτισμές μας σε αντιπαράθεση και σε αντίθεση μεταξύ, του, μεταξύ τους. Μπορέσαμε όμως να βρούμε μια συμπληρωματικότητα με πνεύμα ανθρωπισμού και με ε, ε, τάση αταλάντευτη προς την ελευθερία οι ευρωπαϊκές δυνάμεις απίκησαν την Αφρική και αυτό ήταν ένα αμφιλεγόμενο σημείο αναμφισβήτητα στην κοινή μας ιστορική διαδρομή. Ναι, έχει υπάρξει καταπίεση, εκμετάλλευση, υποδούλωση, κατάκτηση, ακόμα και δουλεία. Ε, πράξεις αποτρόπες ε, σε βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ίχνη από αυτές τις πράξεις δεν θα εξαφανιστούν τόσο εύκολα. Και αυτό το έχουν απαθανατήσει διάσημοι ε, ποιητέ, διανοούμενοι, συγγραφείς, Ευρωπαίοι, Αφρικανοί έχουν ερμηνεύσει και έχουν διερευνήσει όλες αυτές τις ε, σκοτεινές σελίδες της ιστορίας μας. και έχει, ε, η διαδικασία απίκησης έχει αποτελέσει λαμπρό παράδειγμα ελευθερίας και πορείας προς το μέλλον. Έχουν υπάρξει επαρκή παραδείγματα έτσι ώστε τέτοια, τέτοιες πράξεις να μην επαναληφθούν πια παρόλα αυτά δεν ήρθα σήμερα για να αναζωπυρώσω σπισμένες φωτιές και για να, ε, ε, να μετακινήσω το μαχαίρι μέσα στην πληγή έτσι ώστε να την κάνω να αιμορραγήσει ξανά. Αντιθέτως, θέλησα ως εισαγωγική παρατήρηση στην παρέμβαση μου αυτή να υπογραμμίσω τον απαράγραπτο χαρακτήρα των ε, πληγών που έχουν υπάρξει, των τραυματισμών που ε, θα υπάρχουν για πάντα στο συλλογικό υποσυνείδητο των αφρικανικών λαών. Η ιστορία των σχέσεών μας δεν ήταν όμως μόνο θυελώδης και σκοτεινή. Ευτυχώς είναι και μια ιστορία φωτός και γόνιμων ανταλλαγών, γόνιμων επιρροών αμοιβαίων σε πολιτιστικό και πολιτισμικό επίπεδο που μας εμπλούτησαν, που μας έδωσαν νέα πνοή αμφότερους και που μας χειραφέτησαν. Είναι μια συνάντηση η οποία ε, από τον έναν αιώνα στον άλλον οδήγησε σε ένα μοίρασμα ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς της δικής σας και της δικής μας. Κυρίες και κύριοι, το δεθνές περιβάλλον ανασυγκροτείται και αναδιαμορφώνεται με εξαιρετική ταχύτητα. Αναδύονται νέες δυνάμεις και ψάχνουν να βρουν τη θέση που τους αναλογεί σε έναν κόσμο με πολλούς πόλους. Νέες προκλήσεις υψώνονται μπροστά μας, νέα διακυβεύματα και οι βιώσιμες λύσεις θα επιτευχθούν μόνο όταν η δράση είναι συλλογική και αλληλέγγυα. Σε αυτή την αναδιαμορφώση ενός γεωστρατηγικού σύμπαντου που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή και η Αφρική, η Ευρώπη και η Αφρική ε, φαίνεται ότι τάσσονται ε, η μία δίπλα στην άλλη. Έχουν διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές αξίες. Υπάρχει γεωγραφική εγκύτητα και γι' αυτό η μία ήπειρος συμπληρώνει την άλλη. και θα πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση με ισχύ και λογική για να ανθίσει η εταιρική μας σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης θα πρέπει τη συνεργασία να τη στηρίξουμε σε στέρεες αρχές με πολυδιάστατη προσέγγιση, με όραμα, ε, με φιλοδοξία και με επεκτατικές ε, τάσεις ο αμοιβαίος σεβασμός, η ελευθερία και η αλληλεγγύη είναι τα αναπόδραστα βήματα για μια σχέση στέρεα, αμοιβαία εποφελή ε, που θα επιβιώσει και θα αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου. Έχουμε μια φιλόδοξη ημερήσια διάταξη, ένα φιλόδοξο πολιτικό πρόγραμμα για τα 50 επόμενα χρόνια, για την ολοκλήρωση της Αφρικανικής Υπήρου, με, σε συνθήκες ευημερίας και ειρήνης. Είναι μια πολιτική φιλοδοξία και σε αυτήν ε, κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει η στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης και φέτος ε, έχουμε τη δέκατη επέτειο. Έχουμε λοιπόν τους κατάλληλους δείκτες για την μελλοντική μας πορεία και για τη στρατηγική μας εταιρική σχέση. Η Αφρική ήταν και παραμένει το σκηνικό πολλών συγκρούσεων, θανατηφόρων και θανάσιμων ε, στο, στην περιοχή του Σαχέλ, ε, στην περιοχή της λίμνης του Τσάντ, στην κεντρική Αφρική. Παρόλα αυτά υπάρχουν απτά στοιχεία για την ανασυγκρότηση της αφρικανικής Υπήρου. Ο ορυκτός πλούτος, ο θαλάσσιος και αλλιευτικός πλούτος, η ζωντάνια, η ζωτικότητα του πληθυσμού που είναι κατά κύριο λόγο ε, σε νεαρή ηλικία, η χρηστή διακυβέρνηση με το θάρρος και την αποφασιστικότητα της αφρικανικής πολιτικής ηγεσίας η εξάλληψη των τελωνιακών εμποδίων, οι καινοτόμες τεχνικές στη γεωργία και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η καινοτομία στις υπηρεσίες, όλα αυτά είναι κινητήριοι μοχλή για την αναγέννηση της Αφρικανικής Υπήρου. Έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλούς και αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί και να καταπολεμήσουμε ανελαίητα τη διασπάθηση των πόρων, την υπεξαίρεση των πόρων, τη διαφθορά και γι' αυτό βασική προτεραιότητα για εμάς είναι η δημιουργία και η χρήση των κατάλληλων εργαλείων που θα έχουν εγκριθεί σε θεσμικό επίπεδο και από την Αφρικανική Ένωση και από τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε όλοι να τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Η μεταρρύθμιση της Αφρικανικής Ένωσης αποφασίστηκε στη Σύνοδο του Ιανουαρίου του 2017 και αυτό είναι μια ευκαιρία για την αναγέννησή μας ούτως ώστε εμείς να έχουμε τα ενία ε, της οργάνωσής μας, του ε, οργανισμού που έχουμε διαμορφώσει και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτές τις θετικές τάσεις που, έχουν ήδη διαφανεί στον ορίζοντα. Στόχος μας είναι να εξαλείψουμε τα κοινωνικά δράματα που μαστίζουν την Αφρική λόγω ε, ξηρασίας, λόγω λοιμού, λόγω ένοπλων συγκρούσεων και καταστρατηγήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλες αυτές οι συγκρούσεις και οι, κρου... και κρίσεις θέτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ζητούμενο της ειρήνης και της ασφάλειας στις πρώτες θέσεις του καταλόγου των προτεραιοτήτων μας με αποφασιστικότητα θα δράσουμε και για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, τον τζιχαντισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση. Είναι μια μόνιμη και σταθερή δέσμευσή μας υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας και οι προσπάθειές μας είναι ακούραστες, κοπιώδεις για να προλάβουμε, για να διαχειριστούμε και για να ανασυγκροτήσουμε. στηρίζουμε και χαιρόμαστε ε, για την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον αγώνα. Κυρίες και κύριοι, όλες οι μελέτες, οι σημερινές και οι πρόπτικες δείχνουν ότι η Αφρική είναι η, περιοχή του κόσμου που υποφέρει περισσότερο από την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και από την κλιματική αλλαγή. Καταστροφικές είναι οι επιπτώσεις στη Φλωρίδα και στη Πανίδα. επιπτώσεις που ε, καθιστούν ε, περιοχές ολάκερες ε, στην Ήπειρό μας αβίωτες. Η Αφρική είναι αυτός που ρηπαίνει λιγότερο τον πλανήτη και αυτός που υποφέρει περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Η Αφρική παίρνει ελάχιστο ποσό και ποσοστό των διεθνών θυσιών που καταβάλλονται ε, για την ε, καταπολέμηση των ε, κλιματικών αλλαγών. Είναι ένα θέμα που σχετίζεται με την τυρική μας σχέση και θα πρέπει να εξεταστεί καλύτερα, να γίνει αντικείμενο καλύτερης διαχείρισης και να του δοθεί υψηλότερη προτεραιότητα. Είναι ένα προαπαιτούμενο αυτό, μια απέτηση. Θα πρέπει να ανοίξουν μεγάλοι διάδρομοι ε, στο, για το ιδιωτικό τομέα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί το εμπόριο μεταξύ των δύο υπήρων έχει ανέβει, έχει αυξηθεί κατά 50 200 δις ευρώ ετησίως επενδύονται στην Αφρικανική Ήπειρο. Οι επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, κοινωνική και οικονομική ευημερία. Επομένως έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν και θα πρέπει να τους δοθεί ε, πρώτη προτεραιότητα στις πολιτικές μας για τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις. Η οικονομική διακυβέρνηση που ε, υιοθετούμε μας κάνουν να στρέφουμε την προσοχή μας προς τις ε, ελεύθερες συναλλαγές και θα πρέπει οι λογικές ιδέες επενδυτών του ιδιωτικού τομέα να δρομολογούνται Μιλούμε για ένα νέο σχέδιο Marshall για την Αφρική και στη Σύνοδο G20 είχαμε την ευκαιρία αυτά να τα εξηγήσουμε. Η Αφρικανική νεολαία προσωπεί ε, ένα ποσοστό στον παγκόσμιο πληθυσμό που ξεπερνά το 60% και οι γυναίκες είναι άνω του 50% της αφρικανικής ε, οι γυναίκες είναι άνω το 50% του αφρικανικού πληθυσμού. Όλα αυτά είναι μελήματά μας και τροφοδετούν τα προγράμματα που εφαρμόζουμε. Το θέμα της μετανάστευσης είναι πολύ σημαντικό. Μεταναστεύουν νέοι Αφρικανοί στην Ευρώπη και αυτό είναι μια διτή πρόκληση. Χωρίς προετοιμασία ε, υπάρχουν χώρες που ε, βιώνουν την ε, μαζική και αθρώα προσέλευση μεταναστών χωρίς κατάλληλη προετοιμασία, επαναλαμβάνω. Θα πρέπει να επανεφεύρουμε για την νεολαία μας ένα καλύτερο μέλλον εντός της Αφρικανικής Υπήρου. Και άρα η εταιρική μας σχέση Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δράσει προς αυτή την κατεύθυνση. Με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Η Αφρικανική η Διασπορά είναι η έκτη διάσταση της Αφρικής μετά από την βόρεια, την νότια, την κεντρική, τη δυτική και την ανατολική συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ε, Υπήρου και οικονομικά και σε επίπεδο διανόησης και σκέψης. Επέμεινα κυρίες και κύριοι σε αυτά τα οποία είπα στην έννοια της εταιρικότητας, στην έννοια της συνεργασίας. Νομίζω ότι λόγω των κοινών συμφερόντων πρέπει να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό και χαίρομαι που με ακούτε. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ εγκάρδια απέναντί σας και να μην κρύψω τα πράγματα, να μην αποκρύψω μάλλον τα πράγματα γιατί από τη μία θα πρέπει να συνδυάσουμε τον καθολικό χαρακτήρα της εταιρικής μας σχέσης και από την άλλη τον σχετικό χαρακτήρα αυτής της σχέσης. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, υπάρχουν αποχρώσεις διαφορετικές για να μην πω διαφωνίες. Δεν είναι θέμα πολιτικής φιλοσοφίας, δεν είναι θέμα ιδεολογίας επί τη βάση μια συγκεκριμένη ιδεολογία οποία για την οποία με επέλεξαν οι αρχηγοί των Αφρικανικών κρατών. Εγώ πιστεύω στον διάλογο, πιστεύω στην αναζήτηση της συνένεσης, στην αμοιβαία ανακάλυψη, στην συνεργασία, στην αλληλεγγύη ανάμεσα στις θρησκείες και τους πολιτισμούς. Ε, είμαι κατά της κατασκευής τείχων ε, για να, προστατεύει, να προστατεύεται ο ένας από τον άλλο, αλλά πρέπει να υπάρξουν κοινέ προσπάθειες συνεργασίας και κατανόησης. Πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε γέφυρες, έτσι θα μπορέσουμε να αποδεχθούμε την διαφορετικότητα του καθενός. Η πολλαπλότητά μας είναι αν θέλετε η ουσία του δυναμισμού μας και θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας. Θα είναι πραγματικά απαράδεκτο για λόγους διπλωματικής αυρότητας να αποφύγουμε και να αποκρύψουμε την διαφορετικότητά μας. Ε, τα θέματα σαν παράδειγμα της διεθνούς ποινική δικαιοσύνης και της καθολικής δικαιοδοσίας, της σχέσεις ανάμεσα στην δικαιοσύνη, την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Πολλές φορές αυτό το οποίο ακούμε σχετικά με την Αφρική είναι στα αφρικανικά προβλήματα αφρικανικές λύσεις. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν άλοθη για πολιτικούς λόγους. Η επικαιρότητα μας δείχνει ότι τα προβλήματα είναι σοβαρά. Χαίρομαι επίσης για την αναγέννηση της κοινωνίας των πολιτών στην Αφρική και τη συμμετοχή της τομής της συνεργασίας μας. Ίσως θα μου πείτε ότι λέω πράγματα επιπλέον, ότι φορτώνω πάρα πολύ τις εταιρικές μας σχέσεις. αλλά από την άλλη θα πρέπει να θυμηθούμε αυτό το οποίο είχε πει ο Ιούλιος Φέρνα. Τίποτα το σπουδαίο δεν θα συμβεί αν δεν είναι υπερβολικός ο στόχος τον οποίο έχουμε μπροστά μας. Πρέπει λοιπόν με γενεοδορία αλλά και με επιμονή και εργατικότητα να προωθήσουμε τη σχέση μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως βλέπετε ξεκινάμε να χτίζουμε νέες γέφυρες ανάμεσα στην Αφρικανική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είδατε πώς σας χαιρέτησαν οι συνάδελφοι. Θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι όμως και πραγματιστές. Θα πρέπει να εργαστούμε και νομίζω ότι μαζί με την κυρία Μόγκερίνη που είναι υπεύθυνη για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής θα κάνουμε καλή δουλειά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με τα θέματα της Αφρικής, θα πρέπει να υπάρξουν όμως νέες γέφυρες και σε οικονομικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο μεταφορών. Είναι σαφές ότι πρέπει να συνδεθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών με τα αφρικανικά τα οποία τώρα σχεδιάζεται. Θα πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε μαζί από κοινού. Είμαι αισιόδοξο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και σαφείς σε αυτό το οποίο θέλουμε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της τρομοκρατίας και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της μετανάστευσης αν δεν συνεργαστούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, ισχυροποιήσουμε τους δεσμούς μας. Το λέω πάντα στους Ευρωπαίους φίλους. Θα πρέπει να βλέπουμε την Αφρική όχι με γυαλιά Ευρωπαίου, αλλά με γυαλιά Αφρικανού. Αυτό είναι η πραγματική φιλία η οποία θα χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας. Πάντα λοιπόν θα είστε ευπρόσδεκτος σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ.